Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Bonjour Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλημερίζω και σας ε, καλωσορίζω θερμά στην πρώτη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής. Σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη, να σας ενημερώσω ότι δεν προβλέπεται διερμηνία για όλες τις γλώσσες. Για παράδειγμα, βουλγαρικά, τσεχικά, λετονικά, λιθουανικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά και ουγγρικά δεν προβλέπονται στις σημερινές συνεδρίες. Στις επόμενες συνεδριάσεις ε, θα προσαρμοστούμε στην σύνθεση της Υποεπιτροπής εφόσον αριστικοποιηθεί Πάντως προηγούνται τα τακτικά μέλη για τη διερμηνία. Εξού και αυτή η μικρή παράληψη για κάποιες γλώσσες σήμερα και σας ζητώ συγγνώμη. Η συνεδρίαση αυτή αναμεταδίδεται απευθεία από το κανάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, η συνεδρίαση των συντονιστών αναβάλλεται για τις 3 Σεπτεμβρίου, μια και όλες οι ομάδες δεν έχουν ορίσει ακόμη τους συντονιστές τους. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι, οπότε εγκρίνεται. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Θα επανέλθουμε και στην επόμενη συνεδρίαση. Καταρχήν το απόγευμα της 3ης Σεπτεμβρίου θα έρθει στην Επιτροπή μας ο Πατρίκ Μπελουάρ, Διευθυντής της ε, ε, μικτής ε, οργάνωσης για τον εξοπλισμό, συνεργασίας για τον εξοπλισμό και θα μας μιλήσει για τα προγράμματα εξοπλισμού, τα 400M και Τίγρης κυρίως, αυτά τα δύο που χειρίζεται αυτή η μικρή οργάνωση συνεργασίας για τον εξοπλισμό και στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 3 το απόγευμα, προβλέπεται συνάντηση με την ε, ε, Σουηδική Προεδρία και τον πρέσβη Όλαφ Σκουκ του ΚΟΠΣ. Επίσης ασχοληθούμε και με τις ε, αποστολές που θα πραγματοποιήσουμε. Στην Τυρκουάση εβδομάδα στα τέλη Οκτωβρίου που αφιερώνεται σε αποστολές και επισκέψεις των Επιτροπών θα μπορούσαμε να στείλουμε μία λιγομελή αντιπροσωπεία ε, στις επιχειρήσεις Αταλάντα κατά πολέμηση πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ε, αποστολή αυτή στα πλαίσια της ε, ΚΕΠΑ και ο προκάτοχός μου κ. Γκάου με ενημέρωσε τον προηγούμενο Ιανουάριο είχε πραγματοποιηθεί τέτοια αποστολή στο Νόρσκουτ όπου βρίσκεται και το γενικό επιτελείο της επιχείρησης Αταλάντα. Κατά πάση πιθανότητα στα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους ε, θα στείλουμε αποστολή και στο Κωσυφοπαίδιο για να αξιολογήσουμε την πρόοδο της αποστολής Γιούλεξ που δεν είχε αναπτυχθεί πλήρως μέχρι τον Ιούλιο, αλλά σημειώθηκε εντυπωσιακή πρόοδο στους τελευταίους μήνες, γι' αυτό θα ήταν ενδιαφέρον η υποεπιτροπή μας να μεταβεί επί τόπου και να παρακολουθήσει την πρόοδο της Γιούλεξ. Αλλά αυτό θα το εξετάσουμε στην επόμενη μας συνεδρίαση για να δούμε και τις λεπτομέρειες αυτής της αποστολής. Θέλει κανείς το λόγο. Γιάννες. Πότε θα γίνει η πρώτη αποστολή, το Σεπτέμβριο στην Τουρκία. Όχι, όχι στην Τουρκία, στην Τυρκουάζ εβδομάδα. Τέλη Οκτωβρίου, Τυρκουάζ εβδομάδα. Τέλη Οκτωβρίου, στην Τυρκουάζ εβδομάδα, θα γίνει η αποστολή για την, στην επιχείρηση Αταλάντη, δηλαδή στην ε, επιχείρηση που γίνεται για την πάταξη της πειρατείας στις ομελικές ακτές. Άλλος κανείς? Bien. Nous allons donc euh, passer à, à, au principal objet de cette... Euh, Και περνούμε στα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σημείο 3. Ανακοίνωση Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τη μη διάδοση των πυρηνικών. Ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Και ήταν σκόπιμο να εγκαινιάσουμε τις εργασίες μας με το ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό θέμα. Θα ακούσουμε λοιπόν την ε, παρουσίαση της Επιτροπής για τη μη διάδοση των πυρηνικών και κατόπιν ε, την παρουσίαση της ανακοίνωσης σχετικά με την προστασία κατά των χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών και πυρηνικών όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της μη διάδοσης τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μας εκστρατείας γίνονται βαλιστικές και πυρηνικές δοκιμές από τη Βόρεια Κορέα. Αυτό το θέμα διαπίστωσα ότι άγγιξε ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες και οι πολίτες δεν θα συγχωρούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση αν αμελούσε τόσο στρατηγικό ζήτημα. Και υπάρχει κάτι αντιφατικό εδώ. Αφενός έχουμε Πυρηνικέ δυνάμει όπως τη Ρωσία, τις Ηνωμένε Πολιτείε, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που εξετάζουν πολύ σοβαρά έναν πυρηνικό αφοπλισμό και μάλιστα έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ Ομπάμα και Μετβέντεφ πρόσφατα στην Μόσχα και από την άλλη έχουμε μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη διάδοσης των πυρηνικών μέσω των ειρηνικών και βορειοκορεατικών προγραμμάτων. Λογικό είναι λοιπόν να ασχοληθούμε με σοβαρότητα με τα θέματα αυτά και να μπορέσουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε αξιόπιστες και πολύ επικοδομητικές συζητήσεις. Μην ξεχνάτε και το χρονοδιάγραμμά μας που μας υποχρεώνει να αγγίψουμε στα θέματα αυτά. Γιατί το 2010 προβλέπεται η συνδιάσκεψη αναθεώρησης της ε, συνθήκης της μη διάδοσης των πυρηνικών. Κάτι που θα μας ε, τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γκαρίβα, που είναι Ματάρχης της Γενικής Διεύθυνσης ε, Μεταφορών και Ενέργειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Τα λόγια σας ήταν τέλεια εισαγωγή στο θέμα της μη διάδοσης. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να υπογραμμίσω τις προτεραιότητες της ανακοίνωσης αυτής της Επιτροπής. Καταρχάς, τα τελευταία χρόνια, λόγω της κατάστασης στον τομέα της ενέργειας και της ε, αβεβαιότητας των τιμών ενέργειας ανά τον κόσμο, η πυρηνική ενέργεια έγινε θέμα, ξανά θέμα συζήτησης μετά από πολλά χρόνια παραμερισμού κατά κάποιο τρόπο. Τούτο ενίσχυσε σαφώς το πολιτικό ενδιαφέρον όλων των θεσμών της Ένωσης να αναλάβουν δράση και να συμβάλλουν σε συζητήσεις όπως αυτή για την μη διάδοση. Στην ανακοίνωσή της ε, το 2007 για την στρατηγική αναθεώρηση της ενέργειας είχαμε τονίσει σαν επιτροπή την ε, σημασία της μη διάδοσης ως βασικό εργαλείο για την ειρηνική ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας. Αν δείτε πώς καταμερίζεται η εργασία στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι σαφές ότι η βάση γίνεται με την κοινή εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλειας. Οι βασικέ γραμμέ αυτής είχαν καθοριστεί το 2003 από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Το Συμβούλιο συμπλήρωσε τι οδηγίε αυτέ το 2008 με τι λεγόμενε γραμμέ δράση υλοποίηση ε, τη ε, νέα ε, στρατηγική ασφάλεια. Αυτό είναι που, που είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εξ αρχή Είναι ότι Υπάρχουν μεν αυτές οι βασικές γραμμές, υπάρχουν ωστόσο και κάποια εργαλεία και μέσα που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την υλοποίηση των γραμμών αυτών πολιτικής που διαρθρώνονται με βάση την έννοια των 3S, s ασφάλεια, σταθερότητα και ενέργεια το, και προστασία. Οι πολιτικές αυτές που θα συζητήσουμε περιλαμβάνουν μια σειρά διαστάσεων, ε, προστασία από κινδύνους, καθεστώς εξαγωγών, ε, μέσω των, ε, του κανονισμού διπλής χρήσης που αναθεώθηκε. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν, ότι με βάση την συνθήκη Ευρατόμ υπάρχουν πολλές διαστάσεις του θέματος που, καλύπτουν, που καλύπτονται από εκεί. Φερρυπίν, καθεστώτες εσωτερικής προστασίας και συσχετισμός με ε, και συνεργασία και συσχετισμός των δραστηριοτήτων με την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός του χρόνου, την αναθεώρηση τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την ενίσχυση ενδεχόμενα του καθεστώτος μη διάδοση. Το πρώτο λοιπόν σαφές μήνυμα που περιλαμβάνει η ανακοίνωση τη Επιτροπή, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό η Ένωση να ό,τι και να αποφασίσει να εμφανίζεται με ενιαίο μέτωπο εν, προς τα έξω στις, και στην ε, διάσκεψη αυτή. Ζητούμε λοιπόν στην Επιτροπή να υπάρξει ενίσχυση του συντονισμού των εργασιών όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στον τομέα αυτό. Δεύτερο σημείο. Η διεθνή συνεργασία πρέπει να προχωρήσει σε ένα ενισχυμένο διάλογο με την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μέσω των επιθεωρητών της Ευρατόμ και, και μάλλον και οι επιθεωρητές της Ευρατόμ και οι, επι, οι, επιτροπε, οι επιθεωρητές της ΙΑΕ έχουν μακρά παράδοση ελέγχου και επιθεώρησης και συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό. Πέρυσι ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΕ κ. Μπαραντέη, υπέγραψαν ε, ε, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και Διεθνούς ε, Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Η συνθήκη Ευρατών προβλέπει ότι η συνεργασία με βασικούς πυρηνικούς παραγόντες εξασφαλίζεται μέσω μιας σειράς διμερών συμφωνιών. Κατά παράδοση, είχαμε συμφωνίες με τις προμηθεύτριες χώρες, χώρες που προμηθεύουν πρώτη ύλη, Αυστραλία και Καναδά για παράδειγμα, είχαμε επίσης σχέσεις και με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ τώρα διαπραγματευόμαστε εκ νέου μια συμφωνία με τον Καναδά. Οι συμφωνίες αυτές δεσμεύουν τις δύο πλευρές να τηρούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, να, να σέβονται πλήρως τις προδιαγραφέ τη Διεθνού Επιτροπή Ατομική Ενέργεια και την δέσμευση για ειρηνική και μόνο χρήση τη πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει και μια τρίτη παρατήρηση, ένα τρίτο σημείο που συζητείται εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα σε παγκόσμιο πλαίσιο και συσχετίζει το θέμα της του εμπλουτισμού που είναι το πιο πιθανό για διάδοση κομμάτι της πολιτικής, ε, ε, της πυρηνικής πολιτικής, προσπαθώντας να, εξασφαλίσει, να εξασφαλίσουν ότι οι χώρες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς δεν επενδύουν στην τεχνολογία αυτή παρά μόνο αν έχουν σαφές οικονομικό συμφέρον. Δύο πράγματα λοιπόν. Πώς εξασφαλίζουμε ότι η προμήθεια πυρηνικού υλικού χορηγείται στις χώρες εκείνες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Δεν υπήρχε ποτέ έλλειψη πρώτης ύλη στον κόσμο. Είναι σαφές ωστόσο ότι αν επεκταθεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ε, σε μια σειρά χωρών, θα τεθεί το ερώτημα πόσο για οικονομικούς λόγους υλικό θα χρειαστεί οι χώρες αυτές να εμπλουτίσουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να θέσουμε σαν Ένωση μια σειρά ερωτημάτων. Τρεις βασικά ερωτήσεις. Πρώτον, τι κάνουμε με τις χώρες που δεν μετέχουν στο καθεστώς μη διάδοσης. Δεύτερον, τι γίνεται με τις χώρες, είπατε κάποιες εσείς, που μετέχουν μεν στο καθεστώς μη διάδοσης, δεν παρέχουν όμως στην διεθνή κοινότητα επαρκή εγγύηση ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Και τρίτον, χώρες που δεν ανήκουν ή ανήκουν στη, στο καθεστώς μη διάδοσης, πλην όμως θέλουν να βγουν από το καθεστώς αυτό. Αυτά κύριε Πρόεδρε είναι τα βασικά ερωτήματα που θέτει η παρούσα ανακοίνωση. Συνεψή, συνοψίζοντας, ένα, πώς ενισχύουμε τη συμβολή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στην συνθήκη μη διάδοσης και στην αναθεώρησή της. Δεύτερον, πώς επεκτείνουμε, αν πρέπει να επεκτείνουμε την συνεργασία με τις βασικές αναδυόμενες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο. Και τρίτον, πώς συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας τράπεζας πυρηνικού χημικών υλικών και ενός συστήματος παγκόσμιας μη διάδοσης. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο. Η κυρία Νέιτς πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι καλύτερο να ακούσουμε και το Συμβούλιο, μήπως δεν προβλέπετε σε αυτό το στάδιο. Δεν προβλεπόταν. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό είναι άκρο σημαντικό. Εν ώψη και της επικείμενης αναθεώρησης, μάλιστα, της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, το 2005 εξετάσαμε την προηγούμενη αναθεώρηση αυτής της μη διάδοσης, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τότε όμως ε, δεν είχαμε καμία επίδραση στις συζητήσεις ε, της Νέας Υόρκης, γιατί τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανίκανη να συντονιστεί και να εκφέρει ενιαία γνώμη στη συνδιάσκεψη της Νέας Υόρκης. Αν θυμάμαι και πάλι καλά, υπήρχαν αγεφύρωτες τότε διαφορές μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων, των χωρών μελών που είχαν πυρηνικά όπλα και των υπολείπων. Δεν μπορούσαν αυτές οι δύο κατηγορίες κρατών να συμφωνήσουν σε μια κοινή προσέγγιση ε, υπέρ ενός πυρηνικού αφοπλισμού. Εξού και γεφύρωτες διαφορές και η έλλειψη συμφωνίας. Και μάλιστα αυτό συνέβη επί κυβέρνησης Δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία εκ μέρου των Αμερικανών τότε για πυρηνικό αφοπλισμό, για να μην πω ότι ήταν ανύπαρκτη οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση. Οπότε θα είναι σημαντική η διαλύθος αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Πώ θα καταφέρουν τα κράτη-μέλη στη διάσκεψη του 2010 να επεξεργαστούν μια κοινή προσέγγιση και θέση υπέρ της μη διάδοση. Και μάλιστα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής σαφώ και ρητά μας ε, παρουσίασε τις ε, βασικές προκλήσεις για το πώς θα προσεγγίσουμε τις χώρες που δεν έχουν προσυπογράψει αυτή την συνθήκη, άλλες που την έχουν υπογράψει αλλά παρόλα αυτά δεν εξασφαλίζουν ε, κατάλληλο έλεγχο και επίβλεψη, εποπτεία και τέλος πώς θα προσεγγίσουμε τις χώρες που είναι συμβαλόμενα μέρη της συνθήκης αλλά θέλουν να αποχωρήσουν από αυτή. Όλα αυτά βέβαια τα θέματα αναμειγνύονται και με το ζήτημα της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, της μη Ή τι θα γίνει με την πρόταση ίδρυσης μιας τράπεζας πυρηνικών καυσίμων που θα προωθήσει τις ειρηνικές, μη στρατιωτικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας. Και κατά πόσο μια τέτοια τράπεζα θα εξασφαλίσει στις χώρες που το επιθυμούν προμήθεια τέτοιων καυσίμων, χωρίς όμως να πολλαπλασιάζονται οι εγκαταστάσεις για τον εμπλουτισμό του ουρανίου με τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Ελπίζω στην υποπιτροπή μας να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και εκεί η βασική μας προσέγγιση είναι ότι και η πλειοψηφία της Υποεπιτροπής αλλά και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ μιας περαιτέρω ε, περικοπής και περιορισμού των ε, πυρηνικών όπλων και μάλιστα μερικοί είμαστε υπέρ της ε, απόλυτης εξάλληψης των πυρηνικών. Βέβαια, μια τέτοια θέση πολύ κατηγορηματική δημιουργεί προβλήματα στους υπηκόους ε, προσώπους χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα και δεν θέλουν να τα θυσιάσουν. Αυτή είναι πολύ σημαντική πρόκληση λοιπόν και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί εθελοτυφλώτες δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Καλύτερα λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο, κατάματα και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση. Κάτι που περιέπλεξε ακόμη περισσότερο το όλο θέμα και λυπούμε που επανέρχομαι είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση τον ΗΠΑ αντιμετώπισε διαφορετικά τις χώρες που δεν ήταν συμβαλόμενα μέρη της ε, συνθήκης μη διάδοσης, ιδιαίτερα την Ινδία, το Πακιστάν και για να μην αναφέρω μια τρίτη χώρα που επίσης ε, ε, χωρίς ένα συμβαλώμενο μέρος θεωρείται ότι έχει πυρηνικό όπλο. Από άλλες χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη όπως το Ιράν. Υπήρξε διαφοροποιημένη μεταχείριση λοιπόν και αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλιώ δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την μορφή και την ε, υπόνοια ότι χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Γιατί καλές συμφωνίες με την Ινδία και ο εφοδιασμός της Ινδίας με τα υλικά που χρειάζεται και τα καύσιμα για να προωθήσει την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και ταυτόχρονα θέτεται τελείως διαφορετική προσέγγιση προς άλλες χώρες. Βέβαια, στην νέα κοινοβουλευτική θητεία αυτή είναι η πρώτη μας ομιλία, οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε από τώρα απαντήσεις. Εγώ προσπαθώ να αναλύσω τουλάχιστον την κατάσταση και να μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα τις διάφορες προκλήσεις. Ευχαριστώ. Υπογρα... μια σειρά σημαντικών θεμάτων και θα επανέλθω στο τέλο σε μια σειρά πρωτοβουλειών. κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την λεπτομεριακή εισαγωγή που έκανε και τον ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλει η Επιτροπή για να καταπολεμήσει την, τον πολλαπλασιασμό του πυρηνικού υλικού. Όπως είπε και η κυρία Νέιτς προηγουμένως, η συνθήκη μη διάδοσης πρέπει να είναι πάντα σεβαστή. Αυτό είναι ουσιαστικό και για μας και για τη Δυτική Ευρώπη. Βεβαίως, θέλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Θα θέλαμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Να υπάρξει πλήρης εγκατάλειψη του πυρηνικού όπλου και του σεναρίου του της πρώτης επίθεσης. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση για τη δημιουργία μιας τράπεζας ε, πυρηνικού υλικού, αυτό που, την πρόταση που έκανε η Επιτροπή, υπό τον έλεγχο της Διεθνούς ε, Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Άποψή μου είναι ότι η τράπεζα αυτή, η δομή αυτή, θα έπρεπε να περιλαμβάνει χώρες που είναι ικανές να εμπλουτίσουν το ουράνιο. Προσπάθησα να προετοιμαστώ για τη συνάντηση αυτή και να εξετάσω ποιες είναι οι εμπλεκόμενες χώρες. Ε, Γερμανία, η Ιαπωνία εμπλουτίζουν το ουράνιο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλα τα κράτη που μετέχουν στην τράπεζα αυτή θα έπρεπε να παραδώσουν στην τράπεζα αυτή όλο το υλικό που διαθέτουν. Θα έπρεπε το Ιράν, για παράδειγμα, να εγκαταλείψει κάθε ενδεχόμενο να μπορέσει το ίδιο να εμπλουτίσει ουράνιο. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα στις σκέψεις μας άσχετα με το τι είπε ο Ομπάμα για τη συνέχιση της διαδικασίας αφοπλισμού. Τα πυρηνικά κράτη θέλουν να κρατήσουν τα πυρηνικά τους όπλα, το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο πυρηνικές δυνάμεις, Βρετανία και Γαλλία. Ούτε η μία ούτε η άλλη δεν έχουν αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες για να μειώσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο υπό διεθνή έλεγχο. Το άρθρο Έξι της συνθήκης αφοπλισμού είναι βασικό για να λειτουργήσει η συνθήκη μη διάδοσης. Ποια είναι τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξει την τήρηση των δεσμεύσεων των δεσμεύσεών τη από πλευρά των πυρηνικών δυνάμεων. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, πυρηνικέ δυνάμει, να υποχρεωθούν να υιοθετήσουν μέτρα ριζικού αφοπλισμού πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε, να μειώσουμε τα πυρηνικά όπλα. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και η Γαλλία και η Βρετανία έχουν σαφές πυρηνικό δόγμα που προβλέπουν περιπτώσεις χρησιμοποίησης πυρηνικών όπλων. Εμείς χρειαζόμαστε μια πυρηνική λευκή βίβλο που θα προβλέπει σε ένα ε, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο πώς χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα. Ο Χαβιέ Σολάνα και ο Βρετανός Ρόμπερ Σκουπ προέβλεψαν ότι δεν αποκλείεται η χρήση των πυρηνικών σαν πρώτη, ε, σε πρώτη επίθεση. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πολύ πιο φιλόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξετάσουμε την, την υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων ελέγχου και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι οι πυρηνικές δυνάμεις έχουν μια στρατηγική πρώτης επίθεσης αλλά έναντι τίνων, έναντι των χωρών που δεν είναι πυρηνικά κράτη. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να το ζητήσουμε σήμερα. Ο κύριος Βόμποντα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπε η κυρία Νέιτς στο θέμα δηλαδή της νέας στρατηγικής ε, ή της νέας προσέγγισης της ε, νέας αμερικανικής κυβέρνησης που δεν είναι πια και τόσο νέα θα ήθελα να μάθω πρώτα τι είδους επαφές έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, κυβέρνηση Ομπάμα και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις επαφές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο αρμόδιος για τις επαφές και είναι πολύ σημαντικές και οι απορίες της κυρίας Νέιτς γιατί θα ήθελα να διαβεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου και του υπατοεκπροσώπου με τις ε, επαφές της Επιτροπής. Γιατί υπάρχει και άμεση αρμοδιότητα του Συμβουλίου για θέματα αφοπλισμού αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποιο λόγο εδώ. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι το Συμβούλιο μονοπολεί τις αρμοδιότητες για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Επίσης, ρωτώ και πάλι τι είδους επαφές έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος τις εξασφαλίζει με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρόκειται για νέες δομές ε, επαφών μετά τις αποφάσεις που έβλαβε ο Ομπάμα μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρωσία. Ελήθησαν νέες αποφάσεις εκεί για την πολυμέρεια, για θέματα πυρηνικής ενέργειας. Υπάρχει κάτι ορατό, ή κάτι απτό, σε ό,τι αφορά αυτή τη νέα προσέγγιση. Επίσης, όπως είπε και η προλαλή σας, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι Ήδη από φοιτητή, ο Ομπάμα ήταν ιδιαίτερα στρατευμένο σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού. Και ολόκληρο το επιτελείο του, όλοι του οι σύμβουλοι, προβλέπουν σημαντική πρόοδο σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού. Δεν λέω βέβαια ότι όλα είναι μανιχαϊστικά και απόλυτα, αλλά εγώ ευελπιστώ ότι με τις νέες συνθήκες η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων μπορεί να ενισχυθεί. Και σίγουρα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη σύσφυξη των σχέσεων. Μέχρι στιγμή και η Διεθνή Οργάνωση Ατομική Ενέργεια αλλά και ο Διεθνή Οργανισμό είχαν προβλήματα στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου για τι επαφέ που γίνονται σήμερα μεταξύ ΗΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση. σω και στην επόμενη μα συνεδρίαση θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, προσκαλώντας και εκπρόσωπο της Σουηδικής Προεδρίας. Ο κύριος Ζέμκε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί η ανακοίνωση αυτή είναι πολύ σημαντική και τέτοιου είδους ανακοινώσεις θα έχουμε πολλές παρόμοιες ανακοινώσεις. Θα ήθελα να σας ε, επιστήσω την προσοχή στο σημείο 3 στους ε, βασικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της μη διάδοσης. Γιατί νομίζω ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Έχω λοιπόν διάφορες ερωτήσεις. Αρκούν αυτά τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αναφέρονται πολλά και διάφορα μέσα, αλλά υπάρχει ε, μια πολύ σημαντική πληροφορία στη σελίδα 5. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει για την περίοδο 2007-2013 300 εκατομμύρια ευρώ για το μηχανισμό σταθερότητας για την περιοδο παραλαμβανω επαναλαμβάνω, 2007-2013. Τώρα βρισκόμαστε στα μέσα του 2009. Ερωτώ λοιπόν το εξής. Από αυτό το παχυλό κονδύλιο, ήδη απορροφήθηκαν κάποια ποσά. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα αξιοποίηση αυτών των κονδύλιων, τι βαθμός απορρόφησης υπάρχει και πόσα κονδύλια απομένουν μέχρι τα τέλη του 2013. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σχεδιασμό των δαπανών για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν αν τα 307 εκατομμύρια αρκούν, πόσα έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα, τι έχει απομείνει από το κονδύλιο αυτό και πώς θα αξιοποιηθεί. Και νομίζω ότι για πρακτικούς λόγους το οικονομικό θέμα είναι πολύ σημαντικό. Merci. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι το κύριο πρόβλημα είναι η Κορέα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό τα επόμενα πέντε χρόνια να υπάρξει μια συμφωνία με την Κορέα και αν υπάρξει θα την τηρήσουν αυτοί. Το άλλο θέμα είναι η δαπάνη 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η αναφορά στο κείμενο της ανακοίνωσης επιτροπής. Πού θα, κατα... Πού θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Εγώ φοβάμαι ότι είναι πολλά. Merci. Θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου με όσου τάχθηκαν υπέρ, ανάγκης, ε, υπέρ της ανάγκης ε, του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μέσων και μηχανισμών που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το πυρηνικό ζήτημα και τις ανάγκες συνέπειας των κοινοτικών δράσεων. Ερωτήθηκε ποιε είναι οι αρμοδιότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιε οι αρμοδιότητε του είπα εκπροσώπου. Είναι ερωτήσει που επανέρχονται. Επιπλέον, έχουμε και τη θέση ορισμένων κρατών μελών που έχουν πυρηνικό οπλοστάσιο, είναι πυρηνικέ δυνάμει. και την ε, αντίδραση τους να ενταχθούν σε μια κοινοτική προσέγγιση. Φαίνεται ότι αρνούνται ε, ένα είδος ευρωπαϊκής πειθαρχίας σε θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έθεσε μια σειρά ερωτημάτων, αλλά πριν τα απαντήσουμε θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση των ε, χωρών μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της αναθεώρησης του στρατηγικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Γιατί μέχρι στιγμής το ΝΑΤΟ ακολουθούσε το δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που ήταν αδιαφυσβήτητο. Οπότε δεν έχει νόημα εμείς ε, να επεξεργαζόμαστε ε, ωραίες θεωρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της διάδοσης ή για την πρόθεση του πυρηνικού αφοπλισμού, όταν ταυτόχρονα οι χώρες μας δεν ε, ακολουθούν μια συνεπή θέση και στο ΝΑΤΟ. Πάντως ο κόσμος έχει αλλάξει γιατί φαίνεται ότι όλοι τώρα ε, διεκδικούν και φιλοδοξούν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα. Και ο κίνδυνος της διάδοσης δεν είναι απλός κίνδυνος, είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και ένα θετικό στοιχείο στις εξελίξεις αυτές έχουμε τη νέα κυβέρνηση Ομπάμα που μιλά ρητά για κάτι που μέχρι στιγμής ήταν άρρητο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μιλά για ένα κόσμο παραλλαγμένο από πυρηνικά όπλα για πρώτη φορά η Αμερικανική κυβέρνηση. Συμφωνώ λοιπόν με όσους είπαν ότι χρειαζόμαστε ένα νέο είδο σχέσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί πραγματικά συνεργαστούμε και αν προσυπογράψουμε αυτή τη νέα σκέψη της Αμερικανικής κυβέρνησης, μπορούμε να επιφέρουμε πρόοδο και επίσης θα πρέπει να εθετήσουμε συνεπείς πολιτικές συντονισμένες και στην προετοιμασία της συνδιάσκεψης αναθεώρησης της συνθήκης μη διάδοσης, γιατί στο παρελθόν η δράση μας ήταν καταστροφική και ολέθρια στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2005 και αυτή τη φορά έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα το 2010 και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα υποβάλαμε μια διεξοδική δήλωση με συστάσεις για το θέμα αυτό που είναι επίκαιρη αλλά φυσικά θα πρέπει να έχουμε σωστό συντονισμό με τα κράτη-μέλη και κυρίως τις πυρηνικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα δράσεων και μέσων. Για παράδειγμα, αναφέρονται διάφορες δράσεις στα πλαίσια του PSI ή στα πλαίσια της συνθήκης Ευρατόμ. Το πιο σημαντικό όμως είναι η σχέση μας με τις άλλες χώρες, με τις υπόλοιπες χώρες και κυρίως τις χώρες που φαίνεται να περιφρονούν ή να διαφορούν για τη συνθήκη της μη διάδοσης. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι συνάψαμε εμπορική συμφωνία με την Ινδία, μια συμφωνία που δεν περιλάμβανε ρήτρα πυρηνικών όπλων, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επισημάνει αυτή την έλλειψη στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά έπεσε στο κενό η συστάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η απουσία μια τέτοια ρήτρα από εμπορική συμφωνία δημιουργεί ένα πολύ αρνητικό προηγούμενο. Δεν μπορούμε να θαρρύνουμε την Ινδία να συνεχίζει να περιφρονεί την συνθήκη της μη διάδοσης, όπως έγινε και με την αντίστοιχη συμφωνία που σύνυψε η Ινδία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ούτε με το Ισραήλ επικαλεστήκαμε ουδέποτε το πυρηνικό ζήτημα. Δεν έχουμε καν πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε να παραμερίσουμε τελείως αυτό το θέμα, να το αποσιωπήσουμε. Οπότε Πώς να ζητούμε μια Μέση Ανατολή απαλλαγμένη από πυρηνικά ή να διεκδικούμε ειρήνη μεταξύ Ισραηλών και Παλαιστινίων αν αποσιωπούμε τελείως αυτό το θέμα με ένα Ισραήλ που έχει πυρηνικό όπλο. Και αντιφάσεις υπάρχουν και στην πολιτική μας απέναντι στο Ιράν. Και υπάρχουν θέματα που μας επηρεάζουν άμεσα. Για παράδειγμα, τι θα κάνει η κυβέρνηση Ομπάμα ως προς τους αντιβαλιστικούς πυράβλους στο θέμα της αντιπυραυλικής ασπίδας στη Τσεχία και την Πολωνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνασεκ. Καλημέρα. Είμαι νέο μέλος στο Κοινοβούλιο και πραγματικά Χαίρομαι που ακούω όλους όσους, όσοι μίλησαν μέχρι τώρα για την σημασία του να υπάρχει συνέπεια στο θέμα αυτό και από πλευράς ευρωπαϊκών χωρών και από πλευράς λοιπόν χωρών, ιδιαίτερα γνωρίζοντας πόσο επικίνδυνα είναι τα πυρηνικά όπλα και το γεγονός ότι έχουμε την συνάντηση αυτή λίγες μέρες πριν την επέτειο της πρώτης ατομικής πυρηνικής επίθεσης στη Χειροσύμα είναι σημαντικό. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να γίνει μια τέτοια συζήτηση τώρα. Θα μπορούσα να υποστηρίξω απόλυτα αυτά που είπε η κυρία Νέιτς και για την έλλειψη κοινή προσέγγιση από πλευράς Ένωση. Αυτό είναι, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι ε, πρωταγωνιστής στον κόσμο για την ε, μη διάδοση και την αποπυρηνικοποίηση στον κόσμο. Θα ήθελα να ξέρω και άλλοι συνάδελφοι, ιδίως από τις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα, τη Βρετανία και τη Γαλλία. Στη χώρα σας πιστεύετε ότι υπάρχουν πιθανότητες να επιτευχθεί κάτι τέτοιο γιατί όπω ξέρετε και η συνθήκη μη διάδοση ζητάει και από τι χώρε που έχουν πυρηνικά όπλα να προχωρήσουν σε αποπυρηνοκοποίηση, σε μείωση των πυρηνικών τους, ε, του πυρηνικού τους εξοπλισμού. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι εναντί τρίτων χωρών, του Ιράν και άλλων. Είναι πολύ σημαντικό και τα δικά μα κράτη να προχωρήσουν πρώτα στην αποπυρηνικοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι με τον Ομπάμα παρόντα έχουμε πιθανότητες, πολλές πιθανότητες Ελπίζω, ελπίζω, θεωρώ, ελπίζω περισσότερο παρά θεωρώ, ότι αν ήταν εκεί ε, νωρίτερα, αλλιώ είχαν προχωρήσει τα πράγματα στι ΗΠΑ. Τέλο πάντων, τουλάχιστον στον τομέα των πυρηνικών όπλων. Κάτι που θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή και ο κύριος Φόμποντα είπε ότι ελπίζω να υπάρχει την άλλη φορά και κάποιος και από την, το Συμβούλιο, από τη Συνδική για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξέρω και αυτή τη σκέφτονται και τη σκέφτη η Κομισιόν για την νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Ομπάμα είπε πράγματα που δεν είχε πει ποτέ κανένας πρόεδρος τον είπα πριν. Το ερώτημα είναι μπορεί να υλοποιήσει αυτά που θέλει. Εγώ πιστεύω ότι τα θέλει, αλλά υπάρχουν και άλλα συμφέροντα που μπορεί να του πάνε κόντρα. Θα μπορούσε λοιπόν η Κομισιόν, το Συμβούλιο στο μέλλον να μας πούν πόσο μακριά μπορεί να πάει. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει τις προσπαθειές του. Τελευταία παρατήρηση. Αυτή η τράπεζα πυρηνικών, πυρηνικού υλικού. Θα ήθελα να ξέρω κι εγώ, υπήρξε πρόοδος, αν υπήρξε πόση, πότε μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την παρουσίαση της ανακοίνωσης ε, της Επιτροπής και ο τίτλος αυτός καθεαυτός είναι ενδεικτικός. Μη πυρηνική διάδοση. Μη διάδοση πυρηνικό όπλο. Δεν είναι, δεν περιλαμβάνει στρατηγική, στρατιωτικής παρέμβασης, ε, πρώτη αντίδραση, όλα αυτά δεν έχουν θέση συζήτηση εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος σήμερα είναι ένα και λιγότερο ασφαλής. Δεν υπάρχει σαφής αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης. Οι δημοκρατίες που έχουν συνασπιστεί στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μπορούν να υπερασπίσουν εαυτούς με ασφαλή τρόπο, όχι να επιτεθούν, να αμυνθούν. Αυτά όμως δεν είναι αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Τονίζω το εξή. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούμε όλοι με την παράγραφο 4.1 της ανακοίνωσης την ανάγκη ενίσχυσης της υποστήριξης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και των πυρηνικών διασφαλίσεων. Ήδη εδώ πρέπει να υπάρχει συνένεση μεταξύ όλων των κρατών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θέλω να θέσω το ερώτημα που μου ήρθε στο μυαλό αμέσως. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της μη διάδοσης έναντι χωρών που είναι συμβαλόμενα μέρη αλλά δεν προσφέρουν επαρκής διασφαλίσεις υλοποίησης και εφαρμογής της συνθήκης. Ιράν, π.χ. Δεν αναφέρεται βέβαια ρητά η χώρα αυτή. Πολιτικά ε, δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του κόσμου και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΙΕ. Το ζήτημα που τίθεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσει παραπέρα από τις δυνατότητες που έχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας με την Κίνα και τη Ρωσία. Μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων προς το Ιράν. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάναμε εάν συμφωνούσαν η Κίνα και η Ρωσία μαζί μας. Μια τελευταία παρατήρηση. Αναφερθήκαν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μέσα στα πλαίσια του μέσου σταθερότητα και αναφέρθηκε το θέμα της μείωσης ε, του πυρηνικού αφαπλισμού. Και σε σχέση με τις ε, χώρες ε, τέως μέλη της Σοβιετικής Ένωσης υπάρχει ένα πρόβλημα κατά με ότι χρήματα που είχε στη Διαθήκη η Ρωσία στο παρελθόν για πλοία παραδείγματος χάρη που κινούνται για, με, με, με πυρηνική ενέργεια κλπ. Αυτά τα χρήματα τα επέστρεψε η Ρωσία, δεν τα χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα να διαθέτουμε εμείς χρήματα και να μην χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε τέτοια περίπτωση. Ε, να μας πει η Κομισιόν τι θα κάνουμε. Επιστρέφω τα χρήματα, εντάξει, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλους λόγους. Αλλά από την άλλη μεριά ο σκοπός για τον οποίο το είχαμε διαθέσει δεν πληρούνται. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριο Σφαμπάλη. In addition to uh, the comments of my colleague uh, I would like to raise... Θα ήθελα εγώ να θέσω δύο θέματα, παρακαλώ. Κατά πόσον σήμερα μπορούμε να προβλέψουμε κατά πόσον η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία είναι έτοιμες να ακολουθήσουν μια κοινή θέση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή παραμένουν στη θέση τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ ως μόνιμα μέλη. Λοιπόν, θέλουν να μείνουν εκεί, θέλουν να έχουν ένα κοινό μέτωπο με τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε το χρόνο των δυνατών. Το άλλο είναι ότι αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στους ε, στους κρατικούς αν θέλετε παράγοντες το πιο σημαντικό είναι όμως οι μη κρατικοί παράγοντες επιστήμονες που προσφέρουν τις γνώσεις τους σε εκείνο που πιο πολλά, οργανωμένο έγκριμα κλπ. Αυτοί οι μη κρατικοί παράγοντες θα πρέπει κάπως να συμπεριληφθούν στη στρατηγική μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε όλοι εμείς που είμαστε καινούργοι εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίσουμε το μέγεθος του και τις επιτροπές του. Πρέπει να αλλάξει λέει κανένα αυτό που θέλει να πει όταν έχει το λόγο. Θα ήθελα καταρχήν να εγκομιάζω τον εκπρόσωπο της Εκτελεστικής Επιτροπής για την πολύ διαφανή και απλή παρουσίαση που μας έκανε εισαγωγικά. Μου φάνηκε αυτό πάρα πολύ ενθαρρυντικό σε αυτή η πρώτη συνεδρίαση. Επίσης, θεωρώ ότι τα έγγραφα που πήραμε είναι πολύ χρήσιμα για το πρώτο αυτό βήμα. Θα παραμείνω σε κάτι που ήθελα εκ σε να πω. Είναι πολύ ενθαρρυντικά να ακούμε τον κύριο Ομπάμα και τους εταίρους του Σιμόσκα για το πώς συνεννοήθηκαν όσον αφορά τους περιορισμούς, τον αυτοπεριορισμό. στον τομέα των πυρηνικών όπλων, της διάθεσής τους και των αποθεμάτων. Θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι απλώς παρατηρητής αυτών των ε, γεγονότων, αλλά να είναι ενεργός ε, παίκτη επίσης όρης όχι απλώ διαβάζοντα εφημερίδε ε, και βλέποντα την τηλεόραση τι γίνεται, αλλά να διαθέσουμε εμείς ένα σοβαρό και συνεπή διάλογο και να επιμείνουμε στο δικαίωμά μας να ενημερωνόμαστε για κάθε στάδιο των ε, δημιουργουμένων. Το άλλο αφορά κάτι που είπε η κυρία Γκόμες και για το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Ότι αυτός ο πυρηνικός διάλογος ε, στην Μέση Ανατολή του παίζουμε κρυφτούλη κατά κάποιον τρόπο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν θα πρέπει σιγά σιγά να καταστεί πιο διαφανής, πιο υπεύθυνος και να έχουμε καλύτερη πρόσβαση θα πρέπει να έχουμε εκεί μία αποστολή με την φιλοδοξία να είμαστε σοβαροί συμμετέχοντες στο παιχνίδι. Δεν αρκεί να φοβόμαστε πού θα λάβει χώρα ο επόμενος βομβαρδισμός, θα πρέπει να δράσουμε ενεργά στον τομέα. Αυτά με δύο λόγια όσον αφορά την πρώτη μου ομιλία εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σπάσκου. Thank you very much. Well, I think you know... Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, εκτός από το να απαριθμούμε ακριβώς τι θέλουμε και να αναφέρουμε ότι ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα είναι πιο ασφαλής από ένας κόσμος ε, με πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να είμαστε πιο ε, δραστήριοι, πιο ενεργοί στην ε, προσέγγιση μας. Θα πρέπει να αναφερθούμε στο διεθνές περιβάλλον το οποίο ε, δεν απλουστεύει αλλά περιπλέκεται. Και αυτό οδηγεί σε περισσότερα κίνητρα σε χώρες να προστατεύσουν αυτούς με πυρηνικά όπλα. Και αυτή είναι η γενική τάση νομίζω. Ο κόσμος γίνεται πιο πολύπλοκος, οι απειλές είναι πιο πολυάριθμες Και αυτό καθιστά το έργο μας πολύ δύσκολο. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε συνεχώς κατά νου το διεθνές περιβάλλον. Όταν μιλάμε για το Ιράν, μιλάμε για το Ιράν αλλά και για να κίνητρα του Ιράν. Δεν είναι μόνο θέμα να κυριαρχήσουν του μαθενικού κόσμου, αλλά και άλλες χώρες που θεωρούν σημαντικές στην περιοχή όπως το Πακιστάν, όπως η Ινδία έχουν ήδη πυρηνικά όπλα και αυτό είναι ότι η διάδοση οδηγεί σε περισσότερη διάδοση αν θέλετε. Ταυτόχρονα, άμα ζητήσουμε από το ΕΡΑ να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα, εντάξει, αυτό θέλουμε. Οι δικές μας αξίες είναι αυτές και προσπαθούμε να τις κοινοποιήσουμε στους εταίρους μας. ταυτόχρονα. Και εδώ δεν είναι μόνο το Ιράν, και το Ισραήλ και όποια χώρα από την οποία ζητούμε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα. Στην περίπτωση αυτή όμως είμαστε σε θέση να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια. Λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί εδώ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εθνικά κίνητρα, τις εθνικές ανησυχίες της χώρας η οποία οδηγείται στο να έχει πυρηνικά όπλα και να αυξήσει τα πυρηνικά της οπλοστάσια. Αν η και η Ρωσία μείωνα σημαντικά τα οπλοστάσια τους, δεν νομίζω ότι αυτό θα ενθάρρυνε σε άλλες χώρες να το κάνουν. Όχι. Τουναντίον Ορισμένες χώρε θα θεωρήσουν ε, ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να μπουν και εκείνες στο παιχνίδι. Η τελευταία μου παρατήρηση. Να κάνουμε δηλαδή την ανάλυση, όπως σας είπα, να λάβουμε υπόψη και τα εθνικά εκάστοτε κίνητρα. Αν μπορούμε, θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της παραδοσιακής προσέγγισης της μη διάδοσης γιατί καταλήξαμε στην ε, συνθήκη αυτή μη διάδοση κλπ. και το είδο τη διάδοση το οποίο συζητάμε σήμερα. Και κάποιο τον έφερα πολύ καλά. Οι μη κρατικοί παράγοντες. Τι γίνεται με αυτούς. Γιατί έτσι όπως είναι το διεθνές περιβάλλον σήμερα, μη κρατικοί παράγοντες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα όπλα αυτά. Γιατί ξέρετε ότι οι πληροφορίες ε, διαδίδονται, υπάρχουν επιστήμονες που προτείνουν να πουλήσουν τον ε, όποιον προσφέρει τα περισσότερα κλπ. Και τελικά έχω να πω υπάρχουν πάντα διαφορές μεταξύ του να δρώ και του να αντιδρώ. Ευχαριστώ. Κύριο Στράσερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί συγκαλέσατε την Επιτροπή τη συνδρίαση αυτή τη Επιτροπή αμέσω μετά την εκλογή σα και θέσατε αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη. Αυτό δείχνει ότι αυτή η Επιτροπή και γενικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα θέματα τη ε, ασφάλεια. Σαν νέο μέλο τη Επιτροπή αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την θαυμάσια πραγματικά έκθεση, ιδίω για τα τρία συμπεράσματα στα οποία κατέληξε τα οποία θα ήθελα να υποστηρίξω και που θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή μας να προωθήσει την Κομισιόν και το Συμβούλιο να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ιδίως σας αφορά το σημείο 2 Θέλω να επαναλάβω κάτι που είπαν κάποιοι από τους προλαλήσαντες. Η κατάσταση έχει αλλάξει όσον αφορά την ε, τοποθέτηση της αμερικανικής πολιτικής. Ταυτόχρονα όμως ήθελα να προσθέσω ότι η Ευρώπη έχει κάθε ενδιαφέρον να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ρωσία γιατί πραγματικά υπάρχουν ίσως δυνατότητες ε, ελιγμό που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Βάγγελ που είπε ότι δεν έχει κατά νου μόνο μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παρακολουθεί και σχολιάζει, αλλά μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δρά, που αποδεικνύεται πλήρως σε θέση να δράσει. Και θα ήθελα να στηρίξω και το τρίτο σημείο ότι δηλαδή θα πρέπει η Εκκληστική Επιτροπή να πάρει μια εντολή για τη δημιουργία μιας τέτοιας ε, τράπεζας ε, πυρηνικού υλικού. Ε, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ποια είναι τα στάδια στα οποία θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση βάσει των τριών σημείων αυτών. Και τέλο θα ήθελα να ρωτήσω μήπως ακριβώ θέμα αυτή τη πολιτική είναι ε, και σε συμφωνία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στη συνεργασία με τον είπα το εκπρόσωπο, την Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο, αν θα ήταν καλό λέω, να ε, μεταβεί η Επιτροπή μα αυτή ε, στη Μέση Ανατολή, μέσα στα πλαίσια του, της προβληματικής αυτής που εξετάζουμε. Έτσι θα μπορούσαμε πραγματικά να παρουσιάσουμε και προς την κοινή γνώμη ότι αυτός ο τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάτισεν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω προσωπικό εκπρόσωπο του ύπατο εκπροσώπου του κ. Σολώνα, θα ήθελα καταρχήν να σα συγχαρώ για την εκλογή σα στην Προεδρία τη Επιτροπή Αυτή και θα ήθελα επίση να συγχαρώ όλα τα νέα μέλη και τα επανεκλεγμένα μέλη της Επιτροπής και βλέπω επίσης και κάποια μέλη τέως μέλη εθνικών κοινοβουλίων με τους οποίους είχα συνεργαστεί και που ήρθαν εδώ τώρα που ήταν εν μέρη πρόεδροι επιτροπών Άμυνας ή εξωτερικών υποθέσεων εθνικών κοινοβουλίων και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα εκ να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη μελλοντική μας συνεργασία Εξ ονόματος του είπα το εκπρόσωπο σας έστειλα νομίζω κάποιο email με συμπληρωματικές πληροφορίες. Το φυλάδιο ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμπεριλαμβάνει ένα άρθρο του κυρίου Φωνβόκα όπου σας συστήνω να το διαβάσετε. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν κλήθη να μιλήσει για το θέμα αυτό. Γι' αυτό απουσιάζει η Σουηδική Προεδρία. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι προετοιμασμένος να ε, τρυφήσω στην ουσία του θέματος. Αλλά όπως ξέρετε, σήμερα το απόγευμα στις 3 το απόγευμα ο Καρλ Μπίλτε θα είναι παρόν στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Συγγνώμη Εξωτερικών Υποθέσεων. Και βέβαια θα του μεταβιβάσουμε το ενδιαφέρον που έχετε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα είναι παρόν ο Κάλμπιλτ και θα του πούμε αυτά που είπατε και θα το ανακοινώσουμε. Όχι μόνο στην Σουηδική Προεδρία βέβαια, αλλά θα τον δώσουμε και στον το εκπρόσωπο τον κύριο Σολάνα. Όπως είπε ο πρόεδρος εισαγωγικά, ο πρόεδρος της πολιτικής ε, ε Επιτροπής και ε, Πολιτικής Ασφαλείας ΠΕΣΕ e, θα έρθει στις 3 Σεπτεμβρίου εδώ να παρουσιάσει την ε, άποψη της Σουηδικής ε, Προεδρίας για το θέμα αυτό και θα μπορέσετε καλύτερα έτσι να έχετε μια ανταλλαγή απόψεων με τη Σουηδική Προεδρία. Τέλος, όπως ξέρετε, ο υπότος εκπρόσωπος κ. Σολάνα τη ιδιαίτερη σημασία στα θέματα αυτά. Χθες ήταν στο Πακιστάν, σήμερα είναι στο Αφγανιστάν. προς το τοπικό βήμα του ΑΖΙΑΝ και έχει σχολιάσει το θέμα αυτό της μη διάδοσης ε, και γενικά τα πυρηνικά θέματα. Μπορώ να σας προναγγείλω ότι θα είναι παρόν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Η... Πιο νωρίς ήταν αδυνατό να έρθει γιατί ο Σεπτέμβριος είναι πλήρης με συναντήσεις γκύμνης στην Σουηδία και επίσης στο Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά στις 11 η ώρα της 30 Σεπτεμβρίου θα μπορείτε να συζητήσετε τα θέματα αυτών του κ. Σολάνα. Τέλο έχω να σα πω ότι έχω έναν συνάλφο που είναι πολύ γνωστή στην υποεπιτροπή αυτή, την Αναλίζα Σολάνα, που είναι ο προσωπικός, η προσωπική εκπρόσωπο του κ. Σολάνα για το θέμα της διάδεση. Δεν είναι παρούσα, γιατί δεν είχαμε οργανωθεί έτσι, δεν είχαμε προβλέψει τη συνεδρίαση αυτή, αλλά θα μπορέσουμε να δούμε να μπορέσει η κυρία Αναλίζα Τζονέλα να είναι περούσα στην Επιτροπή σας και να σχολιάσει το θέμα αυτό. Και πριν ε, ολοκληρώσω θα ήθελα να πω στην κυρία Λούσινγκ η οποία αναφέρθηκε σε κάποιες δηλώσεις των κυρίων Σολάνα και Ρόμπερ Κούπερ. Ο προκάτοχός σας, ο κύριος Κούπερ, είχε θέσει ακριβώς το ίδιο θέμα και υπήρχαν κάποιες παρεξηγήσεις και με χαρά θα σας αποστείλω την επιστολή που είχε στείλει ο Χαβιέρ Σολάνος στον κύριο Φλούγκερ σε σχέση με την δήλωση του κυρίου Κούπερ. Ε, πρόκειται για μια παρεξήγηση γιατί ήταν εκτός ε, του, της όλης της επιστολής που διαβάστηκα. Θα σας στείλω την επιστολή αυτή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις στις διάφορες ημερομηνίες ε, που θα χρησιμοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε εδώ στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη συνάντηση με τον ε, το εκπρόσωπο τη συνάντηση με την κυρία Τζενέλα, θα συζητήσουμε αυτό. Ο κύριος Πεγιό έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Συνάδελφε πολύ σωστά είπε ο ο συνάδελφο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το κυρίω θέμα εδώ είναι να προετοιμαστούμε για την αναθεώρηση της ε, συνθήκης της μη διάδοση. Και τουλάχιστον αυτή τη φορά να βοηθήσουμε μέσω της Επιτροπής μας στη διαμόρφωση κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ένα θέμα ευρύτατο με πολλά συμφέροντα ισχυρών και μάλιστα δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι γνωστή και φημισμένη για την ισχύ της ε, στην ΚΕΠΑ και την ε, ισχυρή διεθνή της παρουσία. Μερικές φορές είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, αλλά το βασικό δεν είναι να είμαστε δραστήριοι, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε αποτελεσματικοί, όπως είπε και ο προλαλής σας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο δεν θα πρέπει να συγχαίουμε το θέμα της μη διάδοσης με αυτά που είπαν μερικοί για την αποστρατικοποίηση κάποιων κρατών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ακριβής. Μιλά για τους μηχανισμούς που διαθέτουμε, τα μέσα που υπάρχουν και θα πρέπει και να είμαστε ρεαλιστές ως προς τις επαφές που θα έχουμε με χώρες που φιλοδοξούν ε, να, εξοπλιστούν με πυρηνικά. Και θα πρέπει να προσδιορίσουμε κάποιους κοινούς στόχους. Και να έχουμε υπόψη ότι επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ζητήσει τι πυρηνικέ δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήψουν τα πυρηνικά, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν και όλα αυτόματα. Α μην βαφκαλιζόμαστε, γιατί έτσι θα χάσουμε πολύ πιθανό την αξιοπιστία μα σε συζητήσει αν έχουμε τέτοιου στόχου κατά νου. Θα πρέπει λοιπόν στα μέτρα των δυνατοτήτων μα να θέσουμε συγκεκριμένου και ρεαλιστικού στόχου με βάση φυσικά την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από αυτή την άποψη, αν θέλουμε να έχουμε κάποιο βάρος και να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κοινή προσέγγιση, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβάλουμε τις δικές μας προτάσεις και συστάσεις. Και όπω είπε ο κύριος Βόμποντα, θα πρέπει να καταρτήσουμε και ένα χρονοδιάγραμμα ακροάσεων σε συνεργασία με τους Άγγλους και Γάλλους, ώστε μέχρι το τέλος του έτους και στην αρχή του επόμενου να προλάβουμε να διαμορφώσουμε κοινέ θέσεις. Αλλά προσοχή, άλλο μη διάδοση και άλλο αποστρατικοποίηση. Μη διάδοση δεν σημαίνει απόλυτη, απόλυτος φιλερινισμός. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να προσθέσω κάτι σε αυτά που υπόθηκαν. Πιστεύω ότι για τις επερχόμενες συζητήσεις με τον κύριο Σολάνα, την κυρία Τζανέλα και την Προεδρία θα ήταν σκόπιμο να τους ρωτήσουμε σχετικά με το τι συμβαίνει στις πιθανές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόσυρση των αμερικανικών τακτικών όπλων που βρίσκονται στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση Ομπάμα ανέφερε ότι προτίθεται να αποσύρει αυτό το οπλοστάσιο τακτικού εξοπλισμού θα ήταν χρήσιμο να τα βρουν οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς στον τομέα αυτό. Κάτι άλλο σημαντικό. Ποια ήταν η συνέχεια της επιστολής που είχε αποστείλει η Γαλλική Προεδρία στο τέλος της Προεδρίας της. Επιστολή πολύ ενδιαφέρουσα του Πρόεδρου Σαρκοζή που μετά τις δηλώσεις Ομπάμα ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι ήθελε να ξεκινήσει μια στρατηγική συζήτηση για το πυρηνικό ζήτημα. Και το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε τόσα κονδύλια για τις πραγματικές ανάγκες άμυνας. Τελικόπτερα για το Αφγανιστάν, για παράδειγμα, Κάποιοι θα έπρεπε να μην συνεχίζουν να δαπανούν τρελά ποσά σε πυρηνικά όπλα που γνωρίζουν ότι εν τέλει έχουν μόνο ψυχολογική αποτροπή και όχι ουσιαστική στην πράξη. Τρίτον, πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην εμπλοκή της να λάβουμε υπόψη και τους λεγόμενους μη κρατικούς φορείς, non-state actors. Η ερώτηση, σωστό είναι αυτό, αλλά τι γίνεται για την θέσπιση πραγματικού έλεγχου των υπεράκτιων. Αλλιώ ό,τι και να λέμε για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όλων αυτών των μη κρατικών φορέων που απο, βεβαίως αυτοί που αποκτούν πυρηνικά όπλα δεν έχουν και καλές προθέσεις. Αλλά αν μη τι άλλο πρέπει να έχουμε μία συνεπή θέση απέναντι σε τρομοκράτες που θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Τέλος, εν ώψη των διαπραγματεύσεων, ιδίως στα πλαίσια του ΟΗΕ, έχουμε μία εμπειρία εν ώψη της αναθεώρησης της συνθήκης. Πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να προβλέψει η Επιτροπή μας έναν μηχανισμό παρακολούθησης και επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στα άλλα πλαίσια. Έχουμε μια εμπειρία από άλλους τομείς. Η επικοινωνία στο παρελθόν εξ αρχής ήταν χρήσιμη και για τους διαπραγματευτές και για μας. Πιστεύω ότι αν δείξουμε από την αρχή το ενδιαφέρον μας να παρακολουθήσουμε τι κάνουμε, θα κερδίσουμε. Πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρον να έχουμε μια πρώτη επαφή με τους εκπροσώπους της ε, ε, ΕΠΑ. Το ίδιο θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται, τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι στο ΝΑΤΟ ιδιαίτερα με στα πλαίσια τη νέα στρατηγική αναθεώρηση του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριε Ζαλεύσκη. Thank you very much, Mr. Uh, Chairman. I'd like to... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία ορισμένα ζητήματα που έθιξε η κυρία Γκόμες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, αποχώρηση κάποιων τακτικών ε, Αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. Και ιδιαίτερα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη ήταν για μας για χρόνια ολόκληρα ένα εχέγγυο ειρήνης και ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ιδιαίτερα μετά από δηλώσεις ε, Ρώσων αξιωματούχων και υψηλών αξιωματούχων ε, του Ρωσικού στρατού που είπαν ότι ε, ως ανταπάτηση της αντιπυραυλικής ασπίδας θα εγκαταστήσουν ε, πυρηνικού πυράβλους στο Καλίνιγκραντ, στο θύλακα του Καλίνιγκραντ οι Ρώσοι. Βέβαια δεν ακούσαμε τίποτα από τον Ομπάμα ή από Αμερικανούς αξιωματούχους ως προς το θέμα αυτό. Μπορεί εγώ να τα πήρα αλλά τέτοιου είδου δηλώσεις είναι πολύ σημαντικές για μας. Σύμμαχοί μα είναι οι Αμερικανοί και θα πρέπει να προσβλέπουμε σε πιο σφαιρικές ε, και παγκόσμιες λύσεις και για την Ήπειρό μας και θα πρέπει στη διαπραγματεύσεις μας με τη Ρωσική να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, όλες τις ε, κοινοτικές χώρες. και να υποστηρίξουμε τέτοιες ιδέες ε, της Αμερικανικής Διοίκησης αν διατυπωθούν ε, δεν μας εξυπηρετούν. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να συσπηρωθούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μία σφαιρική λύση στο περίπλοκο και πολύπτυχο πρόβλημα της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Euh, και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκαρίμπα, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να απαντήσει σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Ε, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για την πολύ ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χάρη στα διάφορα σχόλια θα επιμείνω σε ορισμένα σημεία της ανακοίνωσης και θα επιχειρήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Καταρχήν, η ανακοίνωση αυτή δεν έχει κανένα, καμία στρατιωτική φιλοδοξία. Θέματα δηλαδή αφοπλισμού ή παρόμοια ζητήματα βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής ανακοίνωσης. Είναι άσχετες με την ανακοίνωση. Μιλούμε για την μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και την πιθανή κατάχρηση αυτής της απόπειρας ειρηνικής χρήσης μη στρατιωτικής χρήσης. οτιδήποτε θέμα στρατιωτικό εκπίπτει της ανακοίνωσης. Τέθηκε ένα ερώτημα για το καταμερισμό των αρμοδιοτήτων. Στην ε, εισαγωγική μου ομιλία είπα ότι αυτό το θέμα εμπίπτει στην ΚΕΠΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν γίνεται πολιτική συζήτηση δεν μπορούν να συμμετέχουν τα διάφορα κοινοτικά θεσμικά όργανα προσπαθώντας να εμπλουτίσουν αυτή τη συζήτηση ή δεν μπορούν να ζητήσουν, ε, όπως ζήτησε και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, μία συνέπεια και ένα συντονισμό στη χρήση των διαθέσιμων μέσων και μηχανισμών προκειμένου να υποστηριχθούν οι διάφορες πτυχές αυτής της πολιτικής. Γιατί η πολιτική υπάρχει, αλλά υπάρχουν και οι μηχανισμοί για την ε, βελτίωση της εφαρμογής της. Υπευλήθησαν και πιο συγκεκριμένα ερωτήματα επί της ανακοινώσεως. Καταρχήν, για τη χρήση του προϋπολογισμού του μέσου σταθερότητας, τα 300 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για την περίοδο 2007-2013. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε θα δημοσιεύσει είτε μόλις δημοσίευσε μια ανακοίνωση για τη χρήση αυτών των πόρων και προβλέπεται για το 2010 η αναθεώρηση του ρυθμού δαπανών των διαφόρων μηχανισμών για να γίνει και ένας απολογισμός και μια αξιολόγηση της χρήσης αυτών των κονδύλιων. Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στην, στο θέμα των μη κρατικών παραγόντων, το ρόλο των επιστημόνων κτλ. Αν διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση θα διαπιστώσετε ότι ήδη από το 1994 βάσει το πρόγραμμα τάσης δόθηκε μεγάλη υποστήριξη σε κάποια, κάποιους τομείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να αποφευθεί τέτοια κατάχρηση ανθρώπινου δυναμικού. Τέτοιου είδους υποστήριξη δηλαδή έχει ήδη ξεκινήσει στο παρελθόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση ίδρυσης Τράπεζας Πυρηνικών Καυσίμων. Το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2008 στη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της ίδρυσης μιας τέτοιας τράπεζας πυρηνικών καυσίμων και θα μπορούσε καταρχήν να συμβάλλει στην ε, ίδρυση αυτή προσφέροντας 25 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τμήμα των κονδυλίων θα προέλθει από κοινέ δράσεις του Συμβουλίου, και ένα άλλο τμήμα των κονδυλίων από την Επιτροπή. Κάτι που μαρτυρεί την ε, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Από ό,τι ξέρω, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για την, για την ίδρυση της τράπεζας αυτής ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Βέβαια, αν επιταχυνθεί η πρόοδος σε ό,τι αφορά την δημιουργία μιας τέτοιας τράπεζας που θα δίνει κίνητρα στις διάφορες χώρες να μην χρησιμοποιήσουν ε, ένα τμήμα του πυρηνικού τους, ε, του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων που θα ενισχύει τη διάδοση αν δοθούν τέτοια ενάυσματα λοιπόν, θα διευκολυνθούν και οι συζητήσεις στη συνδιάσκεψη αναθεώρησης της μη διάδοσης. Τώρα δεν ξέρω αν θα σημειωθεί τέτοια πρόοδος βέβαια και δεν μπορώ εγώ τώρα να προβλέψω τις εξέλιξεις. Νομίζω ότι απάντησα σε μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ ευγενική προσοχή που μου δώσατε. Merci. Ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι ορισμένα θέματα όντως πρέπει να τα συζητήσουμε παρουσία και εκπροσώπων του Συμβουλίου. Και ούτως ή άλλως διαπίστωσε ότι και κάποιοι από εσά θέλουν να είναι παρόν το Συμβούλιο στις επόμενες συνεδριάσεις μας. Χρειάζεται ούτως ή άλλως να αυξηθούν οι επαφές για το θέμα αυτό που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο όπως έδειξαν και οι συζητήσεις εν ώψη και της αναθεώρησης σημειώνω δύο βασικά θέματα πάνω στα οποία πρέπει να εργαστούμε. Πρώτον, την ανάγκη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής θέσης, πολύ το αναφέρατε, μιας θέσης που θα περιλαμβάνει αξιόπιστη και ρεαλιστική θέση όπως ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι και τα ερωτήματα που αφορούν τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ προς διαμόρφωση στρατηγική που πρέπει να διελευκανθεί και να διευκρινιστεί. Πάντως γνωρίζω ότι θα υπάρχουν επαφές και με τις ΗΠΑ και σε πολυμερές επίπεδο για το πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν ιδίω από Σεπτέμβριο και μετά. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να καλέσουμε την κυρία Τζανέλα. Μετά το καλοκαίρι, αλλά σύντομα μετά το καλοκαίρι. Το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά πιεστικό. Θέλουμε μέχρι τον Οκτώβριο να υπάρξει μια κρόαση, το πώς θα το συζητήσουμε βέβαια, επί του ζητήματος, κάτι που όλοι υπογράμμισαν. Θα δουλέψουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό, τόσο ώστε να κλείσουμε τις συζητήσεις πριν το τέλος του έτους. Θα καθορίσουμε ημερομηνίες για τη συνάντηση με την κυρία Τζανέλα και μια ακρόαση Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Και ιδιαίτερα θα λάβουμε υπόψη τις ημερομηνίες που μας αναφέρθηκε 7 Σεπτεμβρίου με τον ε, πρέσβη της Σουηδίας στην, Πολιτική Επιτροπή Πολιτική ε, Ασφάλειας δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει και κάποιοι άλλοι από εσά στι 11.30 να πάμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Α περάσουμε λοιπόν στο επόμενο ζήτημα. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ε, χημικής, βιολογικής, ε, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Άιμαν της Επιτροπής θα μας παρουσιάσει την ανακοίνωση αυτή. Σα δίνω το λόγο, τόσο ώστε να έχουμε και λίγο χρόνο κατόπιν για συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Είναι χαρά για μένα να σας παρουσιάσω το κείμενο που υιοθέτησε στις 20 Ιουνίου Επιτροπή. Εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας της Πυρηνικής Ασφάλειας της αλλά αυτό το κείμενο δεν είναι κείμενο της δικής μου Γενικής Διεύθυνσης, αλλά πολλών. Να αναφέρω και την ε, δουλειά της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι συνάδελφοι από την ΤΡΕΝ, της μεταφορών δηλαδή, για τη μεταφορά των υλικών, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και λοιπόν. Συνεργαστήκαμε μια σειρά άλλων διεθνών οργανώσεων για την προετοιμασία του πακέτου αυτού. Europol, Eurojust, Διεθνής Επιτροπή, Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κλπ. Το κείμενο λοιπόν που έχετε μπροστά σας είναι αποτέλεσμα από πολλούς ειδικού και από ε, μια διαδικασία συνεργασίας και ζητήσεων που ξεκίνησε από τις αρχές του 2008 με συμμετοχή ειδικών από τα κράτη-μέλη. Το 2008 είχαμε γύρω στις 15 συζητήσεις για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα ε, ασφάλειας ε, χειροποίη που να είναι πλήρες, συγκεκριμένο και να καλύπτει όλη την Ευρώπη χωρίς την εμπλοκή όλων αυτών των ειδικών ε, από εθνικό επίπεδο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε προσκομίσει τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Το θέμα τώρα. Το περιεχόμενο και ο τόνος της ανακοίνωσης δεν είναι να δημιουργήσει ανησυχία. Υπάρχει μικρή πιθανότητα να χρησιμοποιούνται υλικά χειδηροποίηση σε πυρηνικέ ε, επιθέσεις. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις ότι η αγορά του υλικού αυτού και η χρήση του σε πυρηνικές ενέργειες είναι δυνατή, δεν είναι πολύ πραγματοποιήσιμη. Είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Αυτή η ευθύνη των κρατών μελών είναι ευθύνη των κρατών μελών, η Επιτροπή ωστόσο έχει ρόλο. Και είναι πολύ πιθανό τα κράτη-μέλη να επηρεαστούν. Η ανάγκη λοιπόν πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Ένωσης είναι χρήσιμη. Το πακέτο που υιοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου περιλαμβάνει και ένα κείμενο εργασίας της Επιτροπής που είναι αποτέλεσμα ε, συνεργασιών με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος και που έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι οι ιδιοκτικές αρχές και οι υγειονομικές αρχές μπορούν να συνεργαστούν όταν έχουν επεισόδιο χιβηροπή. Βλέποντας τα προβλήματα από διαφορετικές διαστάσεις. Προσπαθώντας να δουν σε εθνικό επίπεδο τι θα κάνουμε αυτό. Κάτι πολύ σημαντικό. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε. Δίνοντας μια γενική εικόνα, το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταση της Ένωσης, από την εποχή των επιθέσεων με άνθρακα στι ΗΠΑ είναι σαφέ ότι χρειαζόταν να γίνει περισσότερη δουλειά σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μια σειρά προγραμμάτων που υιοθετήθηκαν. Το καινούριο στην προσέγγιση αυτή είναι ότι εμπλέξαμε όλους τους παράγοντες, όλες τις γενικές διευθύνσεις, έχοντας πετύχει με τον τρόπο αυτό μια συνεκτική αντιμετώπιση του θέματος. Στην ανακοίνωση επίσης θα δείτε μια γενική εικόνα του πώς θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρξει ένα επεισόδιο σήμερα αύριο. Ένα κομμάτι της προσέγγισης αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης έχει πάνω από 130 δράσεις που πρέπει να προχωρήσουν, κάποιες πιο σημαντικές ό,τι αφορά το φόρτο εργασίας από τις άλλες, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι για την εφαρμογή, η υλοποίηση των πόρων, πρέπει να βρείτε κάποια στοιχεία. Κάτι πιο σημαντικό επίσης. Θέλουμε να δημιουργηθεί, προτείνουμε να δημιουργηθεί μια συμβουλευτική επιτροπή χιβιεροπή και να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή και τη διαδικασία αυτής και της συνεργασίας θα παραμείνει στο επίπεδο που θέλουμε να παραμείνει και αυτό θα επιτευχθεί με τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Βλέπετε και κάποια κονδύλια για τη χρηματοδότηση. Γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα τα επόμενα τρία χρόνια για συναφή σχέδια. Υπάρχει βέβαια κονδύ, υπάρχουν κονδύλια και για την έρευνα για την πυρηνική ασφάλεια και τα κονδύλια που αναφέρθηκαν από το εργαλείο στα, από το μέσο σταθερότητα. Δύο λόγια για τις δράσεις αυτές καθεύτερες. Η δομή της περιλαμβάνει τέσσερα βασικά, τέσσερις βασικές, τρεις βασικές διαστάσεις. Πρόληψη, ανταπόκριση και διαπίστωση. Με διάφορα με διάφορες διαστάσεις και στην ανείχνευση και στην ετοιμότητα αντίδραση. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι περιλαμβάνουμε τι θέλουμε να πετύχουμε, να αναπτύξουμε καταλόγους ένωσης ε, χιβυροποίη υλικών. Υπάρχουν πολλοί πίνακες, πολλά, πολλές κατηγορίες, αλλά αυτό που λείπει είναι να έχουμε μία προσέγγιση βάσει του κινδύνου αυτά. Και ότι, οι δράσεις που λαμβάνονται είναι επικεντρωμένε σε θέμα ε, υψηλού κινδύνου χρήση για τις τρομοκρατικέ επιθέσεις. Να δούμε ποια είναι τα επικεντρωμένα υλικά από του διαφόρου καταλόγου και να ξεκινήσουμε με ένα μικρό αριθμό υλικών προσθέτοντα ε, στην πορεία. Επίσης μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την ασφάλεια των ε, υλικών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία τους και την ε, διάθεσή τους ώστε και οι εγκαταστάσει ε, να γίνουν όλο και πιο ασφαλείς. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη με βάση τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων. Ο έλεγχος των ουσιών αυτών είναι σημαντικός και κατά τη χρήση και κατά τη διάθεση και επεξεργασία τους. Γι' αυτό και περιλαμβάνουμε σχετικά εδάφια στο σχέδιο δράσης. Όλες αυτές βέβαια οι δράσεις εξαρτώνται από ε, προσωπικό που ασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα της ασφάλειας, ε, έχει εξοικείωση με τέτοιου είδους υλικά και αυτό ο τομέας της ασφάλειας θα πρέπει να είναι παρόν συνέχεια. Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ύποπτε δράσει, ύποπτε συναλλαγέ, θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένο το προσωπικό με τέτοιου είδου ε, θέματα για να μπορούν ε, να ενημερώνουν τι αρμόδιε αρχέ και να εντοπίζονται οι ένοχοι. Έτσι έχουμε διάφορε δράσεις ό,τι αφορά την ανείχνευση και την ε, καταγγελία ύποπτών συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τη μεταφορά, ήδη υπάρχει σχετική νομοθεσία και αυτό που προσπαθήσαμε ήταν να εξασφαλίσουμε ασφαλή μεταφορά αυτών των υλικών. Και οι εμπειρογνώμονες των μεταφορών θα επιληφθούν αυτόν αυτό το τομέα. Θέλουμε να βελτιώσουμε και την ανταλλαγή των πληροφοριών. Και αυτό το σκοπό έχουν συγκεκριμένε δράσεις για τη βελτίωση της ανταλλαγής των πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά την ανείχνευση, μας ενδιαφέρει μια προσέγγιση με βάση σενάρια για να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε στο θέμα τη προστασία. Να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υλικά προκειμένου να σχεδιαστούν κάποιες τρομοκρατικές ενέργειες και να χρησιμοποιηθούν στις ενέργειες αυτές για να δούμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες ανείχνευσής μας ή πόσο μπορούμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τι γίνεται με την ε, ανείχνευση βιολογικών κινδύνων που είναι πολύ πιο δύσκολη από την ανείχνευση ραδιολογικών ή πυρηνικών υλικών. Επίσης θέλουμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ανείχνευσης σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό ε, Πρόγραμμα Πιστοποίησης. Και όπως είπα και πριν, το θέμα της ανείχνευσης και η ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών, η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμών είναι πολύ σημαντικά θέματα. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα και αντίδραση θα πρέπει να βελτιώσουμε τα εθνικά σχέδια αντίδραση. και οι εθνικοί εμπειρογνώμονε μα λένε ότι υπάρχει δυνατότητα ε, βελτίωση ε, αυτή τη ικανότητας στα διάφορα εθνικά σχέδια. Υπάρχουν όμω και διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών και των εμπειριών που έχουν στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Θέλουμε τα πιο προηγμένα κράτη από την άποψη αυτή να επικουρήσουν τα κράτη που δεν έχουν ακόμη τέτοια μέτρα και να αξιοποιηθούν αυτές οι εμπειρίες. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη δική μας δυνατότητα αντίδρασης και αντιπερισπασμού. Φυσικά θα πρέπει να περιτανεύσει και το πνεύμα της ελεγγύης και αρρωγή των κρατών μελών σε περίπτωση κρίσης. Μιλήσαμε για θέματα εμβολίων, ε, κλινών σε νοσοκομεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά και να υπάρξει αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών μελών για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες κρίσεις. Σε θέματα αντίδρασης, σημαντικό είναι και το θέμα πού θα εντοπιστεί μια απειλή. Και όταν μιλούμε γι' αυτό, μιλούμε και κάποια εργαλεία προσωμείωσης και τις ε, συνέπειες, ε, για παράδειγμα, ενός ραδιενεργού νέφους ή νέφους ε, χημικών ουσιών. Και μάλιστα τέτοιου είδου εργασίε έχει κάνει το κοινό ερευνητικό κέντρο. Πάντω μπορούμε να βελτιώσουμε τα ισχύοντα μοντέλα και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, ότι φορά και πάλι την ετοιμότητα και αντίδραση, θα πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα ερευνών. Βέβαια, ο πρωταρχικός στόχος είναι η διάσωση ζώων και αποφύγει των θυμάτων, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσουμε και ερευνητικά στοιχεία, αποδείξεις, τεκμήρια, για να ανοιχνευτούν τα ίχνη των αυτούργων της ε, τρομοκρατικής επίθεσης. Στο κεφάλαιο οριζόντιες δράσεις υπάρχουν πολλά και διάφορα σημεία. Ίσως η πιο σημαντική είναι η βελτίωση της επαφής με το κοινό, της επικοινωνίας με το κοινό. Και ιδιαίτερα όταν μιλούμε για τέτοια περιστατικά θα πρέπει να ενημερώνεται το κοινό το συντομότερο δυνατό για να αποφευθεί ο πανικός και τα μηνύματα που στέλνονται στο κοινό είναι τα σωστά και μάλιστα υπάρχει ένα δίκτυο αρμοδίων επικοινωνία στα κράτη-μέλη για να εξασφαλιστεί συντονισμό των κρατών μελών σε θέματα αυτά. Οπότε ένα τέτοιο συμβάν έχει λάβει χώρα. Να, δοθεί μια, να υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση και να είναι ενιαίο το μήνυμα προς το κοινό. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται η πρόσβαση σε τέτοιου είδους υλικό χιβιροπή. και όταν μιλούμε για υψηλούς κινδύνους, μιλούμε και για διαδικασίες ε, προστασίας ε, ή αδειοδότησης που θα πρέπει να είναι ενιαίες στα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στη σχετική έρευνα. Ήδη υπάρχουν πολλά προγράμματα τέτοια ερευνητικά και ήδη από τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, έχουν αφιερωθεί 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να δούμε τις σωστέ προτεραιότητε και χάρη στου εμπειρογνώμονες μπορούμε να καθορίσουμε τις προτεραιότητε που θα προωθήσουμε με τα ερευνητικά αυτά κονδύλια. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να ήταν κάπως ε, ακροθυγής αυτή η παρουσίαση, αλλά φαντάζομαι θα σας ε, θα θέσετε πολλέ ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από τρία χρόνια, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, είχα την τιμή και την ευκαιρία να αναλάβω την έκθεση για τις εξωτερικές δράσεις καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας. Και στόχος της γνωμοδότησης αυτής ήταν ε, να δοθεί μια συνέχεια σε μια πρωτοβουλία της Άννας Γκόμες, σε μια ιδέα της Άννας Γκόμες. Μετά τις συζητήσεις που έγιναν ε, για την έκθεση αυτή στις αρμόδιες επιτροπές και στην Ολομέλεια, είχα επαφή με πολλούς συναδέλφους και διάβασα και βιβλιογραφία των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών των μεγαλύτερων κυρίως χωρών, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τότε, ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την 11η ε, Μαρτίου στην ε, Μαδρίτη, διαπίστωσα πώς διάφορες τρομοκρατικές ε, ομάδες και κυκλώματα όπως η Αλκάιντα ενεργούν και διαπίστωσα ότι και το οργανωμένο έγκλημα και τα διεθνή κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν ή προσπαθούν να εξασφαλίσουν τέτοια υλικά. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν τέτοια χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν σε τρομοκρατικές ενέργειες ή στις προσπάθειες εκβιασμού για να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Και μάλιστα μετά την 11η Σεπτεμβρίου το θέμα της πρόληψης και της ανείχνευσης ε, διάφορων τέτοιων υπηρεσιών, πληροφόρησης, μυστικών πληροφοριών και των σωμάτων ασφαλείας των κρατών μελών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αναπτύχθηκαν με ταχύς ρυθμούς. Και μάλιστα, χάρη στην εξέλιξη αυτή, αποτρέψαμε την απόκτηση τέτοιου υλικού από τρομοκρατικές ομάδες, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Πάντως, η ίδια η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση αυτή και η ύπαρξη των κοινωτικών θεσμικών οργάνων δείχνει την ε, ανάγκη αυτής της ε, κοινή προσέγγισης και την αποτελεσματικότητα. Γιατί μεμονωμένα κανένα κράτος από μόνο του θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τέτοιου τους απειλές που είναι περίπλοκες και πολυδιάστατες και η αντίδραση που απαιτούν ε, προϋποθέτει και τεχνολογικές πληροφορίες και μυστικές πληροφορίες αλλά και οικονομικές ε, δυνατότητες που κανένα κρατός μέλος μόνο του δεν θα μπορούσε να τις αναλάβει. Εκεί φάνηκε λοιπόν πόσο αναγκαία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας από τους τομείς που η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδειξε πόσο σημαντική είναι. Φυσικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε πανικό, ούτε να κινδυνολογούμε προκειμένου να θορυβούμε τους πολίτες. Θα πρέπει όμως οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια, να έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι γίνεται. Και όταν υπάρχει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, έτσι εξασφαλίζεται και η ασφάλεια και η ηρεμία των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης ε, εύκολες ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και κοινή δράση. Επαναλαμβάνω ένας από τους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει πόσο επιτακτική ανάγκη συνιστά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τον Λιτζάνες ε, ότι εδώ έχουμε έναν τομέα στον οποίο πραγματικά είναι αναντικατάστατη η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει πραγματικά να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα της Κομισιόν. Το θέμα που τίθεται είναι πότε αυτή η task force κάνει τακτικούς ελέγχους στα κράτη-μέλη για να εξετάσει κατά πόσον τηρούνται οι διατάξεις που έχουν επιβληθεί. Είναι ουσιαστική σημασία σε αυτό, γιατί είδα από την εμπειρία στη χώρα μου ε, ιδίως πούμε και όσον αφορά το θέμα της ε, εφαρμογής ε, των υποχρεώσεων που έχουν ληφθεί μέσα στα πλαίσια της σύμβασης για τα χημικά όπλα, ότι από τη λέξη μέχρι την πράξη υπάρχει τεράστια απόφαση. Και αν δεν υπάρχει κάποιο όργανο, κάποια υπηρεσία που σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρακολουθεί τι γίνεται, δεν γίνονται πολλά. Καμιά φορά οι ίδιοι εμπειρογνώμοντες που έρχονται εδώ ε, αισθάνονται τελείως ανίκανοι να επιβληθούν στις αρχές της χώρας τους. Αυτό γίνεται στη χώρα μου. Είμαι σίγουρη ότι γίνεται και σε άλλες χώρες. Κατά γνώμη λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα τακτικών επιθεωρήσεων στις χώρες. Γιατί πρόκειται για πάρα πολύ δύσκολα ε, θέματα που πρέπει να ελέγχονται. Ναι, μιλάμε πούμε, για εκρηκτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται και από ε, κατασκευαστές κτηρίων. Αν δεν υπάρχει ένας έλεγχος, αυτές οι ουσίες μπορεί εύκολα να πέσουν ε, στα χέρια υπόπτων. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα τακτικών επιθεωρήσεων για να βοηθήσει τους συμπερογνώμοντες. Ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Σκάλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ από πλευρά μου θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα 133 μέτρα από το πρόγραμμα δράσης θα βρισκόμαστε σε ασφάλεια. Αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει εκεί. Αναφέρεται και στην ανακοίνωση αυτή ότι πολλέ από τι αρμοδιότητε είναι ακόμα στα χέρια των κρατών μελών. Αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε, μεν. Απ' την άλλη μεριά όμω σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να δρούμε από κοινού, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες στα τρία κύρια σημεία της εργασίας. Πρόληψη, ανάληψη και αντίδραση. Από τη μια μεριά προσπαθούμε να καταποτολίσουμε τις θερμοκρατικές δράσεις. Έχουμε την Ευρωπόλ, παραδείγματο χάρη. Αλλά η Ευρωπόλ ε, δεν μπορεί παρά να δράσει εφόσον το επιτρέφουν τα κράτη-μέλη. Αν άλλοι πληροφορίε από τα κράτη-μέλη δεν φτάνουν στην Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν έχει μια πλήρη εικόνα πολλά μπορούν ακόμα να γίνουν για τη βελτίωση λόγω και της απειλής δυνάμει που υπάρχει. Για να ξεπεράσω ο στην στενή εθνική οπτική γωνία. Ένα αυτό. Μετά όμως τι γίνεται εάν κάτι πραγματικά συμβεί. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις λεγόμενες best practices, τις άρτησες πρακτικές στα διάφορα κράτη-μέλη, και να δούμε κατά πόσον τα εκάστοτε ε, στάνταρ που υπάρχουν μπορούν να βελτιωθούν και θα πρέπει να υπάρχει μια δικτύωση μεταξύ των κρατών για να μπορέσουν να αντιδράσουν αν πραγματικά γίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι όσον αφορά τις αντιδράσεις στον πολιτικό τομέα θα πρέπει να είναι η ίδια αντίδραση σε περίπτωση δυστυχήματος ή σε περίπτωση επίθεσης. Δηλαδή, εάν υπάρχει ε, μία περίπτωση στην οποία ένα τρένο, παραδείγματος χάρη, ξοραίστηκε γιατί, ε, δεν, ε, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα και χύνεται τέτοιο υλικό στο χώμα, στους δρόμους, θα πρέπει να αναλυφθούν τα ίδια μέτρα όπως στην περίπτωση που πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση θέση. Αυτό γίνεται στο υψηλότερο δυνατό ε, επίπεδο. Είτε το τρένο έχει εκτροχιαστεί, είτε έχει επιτεθεί κάποιος στο κράτος αυτό. Αυτές οι συμφωνίες λοιπόν που προβλέπει η Κομισιόν θα πρέπει να εφαρμοστούν και στην Επιτροπή μας και στις άλλες ε, συναρμόδιες επιτροπές θα πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα μέτρα που προβλέπονται να εφαρμόζονται πραγματικά στα κράτη-μέλη μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Άγκες. Ευχαριστώ. Νέο μέλος είμαι. Μαθαίνω ακόμα και ίσως να κάνω λάθη σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να κάνουμε. Δύο λόγια θέλω να πω για την αλληλεγγύη στην κοινή μας μάχη κατά του φαινόμενου της διάδοσης στην Ευρώπη. Αναφέρω δύο λόγια από το κείμενο που μιλούν σαφώς, θα το διαβάσω στα γαλλικά, γιατί το γαλλικό κείμενο έχω. I have καλεί την Επιτροπή σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της να συνεχίσει τις εργασίες στον τομέα χειροβιπή για, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις ενδιαφερόμενες πλευρές αποφεύγοντας την επικάλυψη για στο εξωτερικό επίπεδο αυτή η επιχειρησιακή δράση έχει τρία επίπεδα, περιλαμβάνει την στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Επιτροπής. Η ερώτησή μου είναι η άποψη της ελεγγύης μεταξύ των κρατών είναι σημαντική για, για μένα. Η ερώτησή μου είναι μέσα στην αλληλεγγύη αυτή εν ώψη της επερχόμενης δουλειάς, πώς θα ενσωματώσουμε τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Στις μετακομμουνιστικές χώρες, για παράδειγμα, όπως ξέρετε από Κύπρο έχουμε από μια τέτοια χώρα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές συνθήκες και πολλά δίκτυα που είναι κληρονομιά του κομμουνισμού, του Σοβιετικού μπλοκ, των μυστικών υπηρεσιών. Τα δίκτυα αυτά παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διάδοση των πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, κυρίως οι σχέσεις ε, των δικτύων αυτών με το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη εξαγωγή ε, πυρηνικού υλικού. Η ερώτησή μου είναι Ξέρω ότι εδώ στην Επιτροπή κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση. Ενώ αυτό που θέτω εγώ είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα. Θα έλεγα υπάρχει δυνατότητα να ενσωματώσουμε στο κοινό ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας και της διάδοσης τις ειδικέ εθνικές συνθήκες και την ύπαρξη εγκληματικών δικτύων σε κάποιες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα πετύχει αν λειτουργήσουμε με βάση την αλληλεγγύη. Και για την αλληλεγγύη αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εθνικές ειδικέ τοπικές συνθήκες. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη των δικτύων αυτών που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες αυτές σε κάποιες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το υλικό που μας μοίρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω όμως ένα αναπάντητο ερώτημα. Η βασική σημασία όλης αυτής της διαδικασίας ε, εξασφάλισης της ε, χημικής, ραδιολογικής, ε, βιολογικής και πυρηνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στην σωστή διάγνωση και τον προσδιορισμό των απειλών που είναι πραγματικές απειλές. Γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να αποτρέψουμε τις απειλές πρώτα θα πρέπει να ξέρουμε με σαφήνεια περί τίνος πρόκειται. Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι για την κατάρτιση αυτής της τεκμηρίωσης ε, ε χρειάστηκε τη βοήθεια πολλών οργάνων, μεταξύ άλλων και της Ευρωπόλ. Δεν ε, κατάλαβα όμως αν με κάποιο τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου και της απειλής, υπάρχουν δυνατότητες τέτοιες συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών και των ιδιαίτερα των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Γιατί κάθε κράτος έχει την κεντρική υπηρεσία πληροφοριών. Και εγώ ε, ξέρω ότι, γιατί ήμουν, ε, υπηρέτησα στο Υπουργείο Άμυνας και ξέρω ότι οι μυστικές υπηρεσίες είναι υπόλογε εκεί. Τι δυνατότητες υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιοποιήσουμε τις γενικές τουλάχιστον εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Γιατί νομίζω ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι η αστυνομία, για παράδειγμα, για τέτοιου είδους θέματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαμπάλεν σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Ζέμκε. Είπε η Επιτροπή ότι η κίνδυνη είναι μικρή. Το υλικό αυτό ωστόσο χαρακτηρίζεται ως υλικό των φτωχών. Εύκολα το μεταφέρεις, εύκολα το, ε, το, το, το, το, το, συλλέγεις. Ε, γι' αυτό θέλω να ξέρω πώς κρίνεται ότι η κίνδυνη είναι χαμηλή. Να ξαναδώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για την θετική απάντηση και ανταπόκριση στην κίνηση της Επιτροπής. Πρώτη ερώτηση. Η Task Force και η υλοποίηση ε, Τη ανακοίνωση μέσω των επιθεωρήσεων. Αυτό ξεπερνάει τα όρια μα. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε εμεί τι επιθεωρήσει αυτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντα κατά μέρο βέβαια του υφιστάμενου ήδη μηχανισμού. Η Task Force έχει στόχο να λειτουργήσει ω συμβουλευτική ομάδα προ ε, την Επιτροπή. Αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι να υπάρχει σύνδεση με τι αρχέ των κρατομελών, ούτω ώστε να μα λένε αυτέ τι γίνεται. Αν δείτε την ανακοίνωση θα διαπιστώσετε ότι θα υπάρξει μια ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράση, που θα περιλαμβάνει και μια επισκόπηση του πώ έχουμε προχωρήσει ό,τι αφορά την εφαρμογή των δράσεων αυτών. Οπότε προφανώ θα χρειαστούμε και την ε, συμβουλή τη ε, Συμβουλευτική Επιτροπή Χιβιεροπή. Ε, για την υλοποίηση του επίπεδου των μελών. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εθνικές ειδικέ καταστάσεις και την ύπαρξη δικτύων. Έχουμε την δυνατότητα και τα εργαλεία υπάρχουν διαθέσιμα μέσω της Europol. Αναφέρθηκε και από κάποιους άλλους βουλευτές στην Europol η εθνική η οι εκπρόσωποι των εθνικών αρχών, η Αξιωματική σύνδεσμοι δηλαδή, ε, που μετέχουν εκεί εξετάζουν τέτοια φαινόμενα διάδοση υλικών και μπορούν να συναφερήσουν ακριβώς τις ειδικές, ε, τις ειδικές εθνικές καταστάσεις. Αυτό κάνουν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι και ανάλογα με τον τομέα στον οποίο είναι εξειδικευμένοι. Το θέμα της ανάλυσης κινδύνου και της εμπλοκής των μυστικών υπηρεσιών επίσης είναι ένα θέμα ε, που απαντάτε εύκολα. Ζητήσαμε την άποψη των μυστικών υπηρεσιών. Πριν όμω έχουμε και στι Βρυξέλλε αυτό το κέντρο αντιμετώπιση κρίσεων που είναι ακριβώ ε, αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα, καλύπτοντα όλου του ε, κινδύνου που αφορούν χειροβιπή. Τα στοιχεία που ζητούμε θα επιβεβαιωθούν και από την υπηρεσία αυτή. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να εμπλοκεί και αυτού του οργανισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε μήπως άλλες παρατηρήσεις. Μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση. Πρόκειται για ένα θέμα βέβαια που θα παρακολουθήσουμε και οπωσδήποτε θα επιστήσουμε την προσοχή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής ε, ε, Δημοσίων Ελευθεριών στο θέμα αυτό για να μπορέσει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση του τόσο σημαντικού θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις, θα ήθελα να σας υποθυμίσω ότι η επόμενη μας συνεδρία είναι στις 3, 3 Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου το πρωί. Θα υπάρχει ένα συντονισμό στην παραμονή. Και σε εκείνους που φεύγουν τώρα, τους εύχομαι καλές